Κυρίσω την ε, επανάληψη τη ε, Συνόδου Ολομέλεια που είχε διακοπεί στι 19 Απριλίου 2018. Τα πρακτικά τη συνεδρία στι 19 Απριλίου ε, έχουν μοιραστεί και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσει θεωρούνται εγκεκριμένα.